Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Συνάδελφοι, φίλοι, ξεκινάει η πρωινή μας συνεδρίαση. Συνεχίζουμε τη σύνοδο. Κυρία η κυρία Μουνίθ έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες το βράδυ, λόγω του ρυθμού εργασιών στην Ολομέλεια, δεν μπόρεσα να αναφερθώ στον Ορλάντο Ζαπάτα, το οποίο Θάνατο είναι πηγή μεγάλη θλίψη για την ισπανική αντιπροσωπεία. Πέθανε μετά από περγία πείνα. Ήταν ο πρώτο φυλακισμένο συνειδήσεως που πέθανε στην Κούβα τα τελευταία 40 χρόνια και ζητούμε την απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων συνειδήσεω, αντίστοιχων συνειδήσεω στην Κούβα. Και στέλνουμε τα συλληπιτήριά μα και στην οικογένειά του και στο λαό τη Κούβα και ελπίζω ότι το θλιβερό αυτό γεγονό ήταν δυνατότητα να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να σκεφτεί τη σχέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Κούβα σε διμερές επίπεδο που θα δημιουργήσει μόνιμο επικοδομητικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίση βάσεω των άλλων συμφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ήταν θέμα διαδικαστικό αυτό που αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό θέμα για να το αναφέρουμε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση της κυρίας Πατράου Νέβες